Η ομάδα του ΑΕΛΚ και των ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ζήτησαν να οριστεί η κυρία Ντίτ Μπάουερ στην Επιτροπή Λίμπε και ο κύριος Έμερ Κοστέλο στην ε, αντιπροσωπεία με την Παλαιστίνη. Εντάξει, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ερχόμαστε λοιπόν Στι συζητήσει επί περιπτώσεων παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη Δημοκρατία και του κράτου δικαίου, πρώτα απ' όλα η θανατική ποινή στη Λευκορωσία, ειδικότερα οι περιπτώσει των Δημήτρη Καβαναβαλάου και Ουλατσισλάου Καβαλίου. Ε, για ένα λεπτό, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Στην αίθουσα αυτή έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την πολιτική κατάσταση στην Λευκορωσία και πολλά ψηφίσματα έχουν υιοθετηθεί για τη χώρα αυτή. Τώρα θα μιλήσουμε για μια συγκεκριμένη πτυχή της πραγματικότητας της ε, Λευκορωσίας που σχετίζεται με την επιβολή της θανατικής ποινής στη χώρα αυτή υποτιθέμενων ε, τρομοκρατών ε, στο μετρό του Μίνσκ που καταδικάστηκαν ε, σε θάνατο. Έχουμε λόγους να αμφισβητούμε την ε, ε, δίκη αυτή και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Και καλούμε τις αρχές της Λευκορωσίας να αναστείλουν την θανατική την εκτέλεση δηλαδή, και να επιβάλλουν ένα γενικό μορατόριο στις εκτελέσεις. Επίσης καλούμε τις αρχές της Λευκορωσίας να σταματήσουν να παρενοχλούν τους ε, ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών και να απελευθερώσουν όλους τους πολιτικούς κρατούμενους. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Το λόγο ο Μιζάλσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Όπως αναφέρθηκε ήδη, δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα αποφασίσουμε ποιος είναι ένοχος και ποιος όχι, αλλά στη διαδικασία ε, διευκρίνησης τούτη συνέβη στην ε, τρομοκρατική ενέργεια στο μετρό του Μόρσκ ε, είναι προφανές ότι πολλά από τα στοιχεία ε, είναι αποτέλεσμα ε, απόσπασης ομολογιών με ε, βασανιστήρια από τους υπόπτους. Δεν είναι ο ρόλος μας να πούμε αν κάποιος είναι ένοχος ή όχι, ε, αλλά μπορούμε να πούμε ε, ή να πούμε αν είναι θανατική ποινή, είναι καλή ή όχι. Αυτό για το οποίο μιλάμε είναι μια σαφή καταδίκη και απόρριψη ε, αυτών των συγκεκριμένων περιπτώσεων θανατικής ποινής Νομίζω ότι πάντα θα πρέπει να είμαστε κατά της θανατικής ποινή σε μη δημοκρατικά, απολυταρχικά και αυταρχικά καθεστώτα. Γιατί η θανατική ποινή είναι ε, πάντοτε ένα ακόμα μέσο κατά των αγώνων του λαού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχάλης η κυρία Γκέριγκερ Εντεμπερκ για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Πέρσι εγκρίναμε τέσσερα ψηφίσματα συνολικά με θέμα την παρενόχληση της ε, κοινωνίας των πολιτών και των υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σήμερα συζητάμε την περίπτωση του Δημήτρη Καναβάλαου και του Λαντίσου Καβάλιου για εικαζόμενη διάπραξη τρομοκρατικών ε, επιθέσεων το 2010 στο μετρό του Μίνσκ. Υπάρχουν ε, πολλές επιφυλάξεις όσον αφορά τη διεξαγωγή της δίκης οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαμορφώνουν γενικά την κοινή γνώμη Ε, αλλά οι ανακρίσεις γίνονται στη βάση βασανισμών, βασανιστήριων. Ε, ε η ενοχή των δύο, αυτών, των δύο αυτών κατηγορουμένων δεν είναι ξεκάθαρη. Ε, γι' αυτό σας, ε, θα πρέπει να αντιδράσουμε για να τεθεί ένα τέλος στην επιβολή θανατικών ποινών. Θα πρέπει να εφαρμοστούν κάποιες κυρώσεις στο καθεστώς της ε, Λευκορωσίας. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ούντεμπεργκ. Η κυρία Λόχ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ενώ παγκοσμίω μειώνεται η επιβολή τη θανατική ποινή, η κυβέρνηση Λευκορωσία ω μοναδική ευρωπαϊκή κυβέρνηση συνεχίζει αυτή την πρακτική. Ο πρόεδρος Λουκασέγκο, ο οποίος αρέσκεται να τονίζει την επιθυμία προσχώρησης τη χώρα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ένωση ε, δεν βλέπει, δεν αναγνωρίζει ότι η επιβολή θανατική ποινή είναι ασύμβατη με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, 400 άνθρωποι ε, εκτελέστηκαν από την θέσπιση θανατικής ποινής. Ε, η στιγμή της εκτέλεσης δεν γνωστοποιείται ούτε καν στα μέλη της οικογένειας. Ενώ τα σώματα των εκτελεσθέντων δεν δίδονται στους συγγενείς τους για ενταφιασμό, ούτε γνωστοποιείται ο τόπος ε, ταφής τους. Και τώρα ο Δημήτρη Καναβάλοφ και ο Λάντισλου Καβάλου θα εκτελεστούν παρόλο που η διεξαγωγή της δίκης δεν ήταν δίκαιη. Οι κανόνες του κράτους δικαίου δεν ε, τηρήθηκαν και τις έναμες τάξεις και πολλά συνηγορούν ότι οι ομολογίες αποσπάστηκαν με βασανιστήρια η θανατική ποινή μπορεί να εκτελεστεί ανα πάσα στιγμή. Γι' αυτό η διεθνή κοινότητα θα πρέπει να ενισχύσει την άσκηση πίεση στην κυβέρνηση του Μίνσκ. Καλούμε μέσω αυτού του δημοψηφίσματο να ανασταλεί η εκτέλεση τη ποινή και να θεσπιστεί ένα μορατόριουμ για την θανατική ποινή έω ότου ε, καταργηθεί πλήρω. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Λόχ Πίλερ. Ακολουθεί ο άνθρωπο κύριος Μαστάλκα για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο καθένας από εμά γνωρίζει την αξία της ανθρώπινης ζωής. Εγώ ως ιατρός γνωρίζω πολύ καλά την αξία της ανθρώπινης ζωής. Συζητούμε για ένα ψήφισμα σε σχέση με την θανατική ποινή για τον Καναβάλιο και τον Καβάλιοφ και το συνδέουμε με το γενναιότερο θέμα τη κατάργησης τη θανατικής ποινή στη Λευκορωσία. Ποια είναι τα γεγονότα. Η θανατική ποινή είναι, ένα, είναι μια ποινή που προβλέπεται στα δίκαιο της Λευκορωσίας για βαριά αδικήματα. Η κυβέρνηση της Λευκορωσίας έχει εξαγγείλει ένα μορατόριο σε σχέση με την επιβολή της θανατικής ποινής. Οι καταδικασθέντες είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν χάρη από τον πρόεδρο. Ένα το έπραξε, ο άλλο όχι. Η τρομοκρατική επίθεση στο μετρό του Μίνσκ ε, δεν ε, ε, ερευνήθηκε μόνο από τις αρχές της Λευκορωσίας, αλλά και από μυστικές υπηρεσίες ευρωπαϊκών χωρών. Ε, πράγματι έγινε τρομοκρατική επίθεση με θανάτους αλλά ε, δεν θέλουμε να καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι, οι καταδικαστέντες ε, χωρίς ε, την ύπαρξη επαρκών αποδεκτικών στοιχείων. Θα ήταν μια επιτυχία να αρθεί η θανατική ποινή σε αυτή τη χώρα και αυτό βάσει του νόμου είναι δυνατόν να γίνει όπως και στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Είμαι σταθερά πεπισμένος ότι χρειαζόμαστε, θα πρέπει να πετήσουμε τουλάχιστον ένα μορατόριο και μια κατάργηση της θανατικής ποινής. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Καστάλκα. Ακολουθεί ο συνάδελφος κύριος Γκερμπράντη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συμφωνήσω με όλους αυτούς οι οποίοι ζήτησαν την αναστολή της εκτέλεσης της θανατικής ποινής στην Λευκορωσία. Η Λευκορωσία έχει εφαρμόσει, έχει εκτελέσει τη θανατική πονή 400 φορές τα τελευταία 9 χρόνια. Συνέχεια βλέπουμε ανθρώπους να φυλακίζονται και να τους επιβάλλονται ποινές βάση υποτιθέμενης επιχειρηματολογίας η οποία προβάλλεται. Όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που ε, είναι τρόφιμοι φυλακών. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά γίνονται επί τη βάση ιδεών. Εμείς έχουμε το μότο του έργο sum». Αν όμως δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί σύμφωνα με την κυβέρνηση αυτή, τότε δεν έχει το δικαίωμα να υπάρχει, να στηρίξουμε το δικαίωμα των ανθρώπων ε, στην ανθρώπινη τους ύπαρξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εξ των πολιτικών ομάδων, καταρχήν ο κύριος Στάσενεκ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προσωπικώς ανησυχώ ιδιαίτερως με την υποβάθμιση ε, της κατάστασης ως προς το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λευκορωσία. Ε, δίδονται αναφορές για βασανισμούς και για απάνθρωπες ε, συνθήκες διαβίωσης των πολιτικών κρατουμένων. Μετά μάλιστα και τις εκλογές. Δύο νέοι φυλακισμένοι έχουν καταδικαστεί σε θάνατο και όλη αυτή η δίκη, η καταδίκη και η διαβίωση του στις φυλακές έχει, βασίζεται σε πάρα πολλά περιστατικά μη δίκαιης δίκαιης γενικότερα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να στηρίζει τις οικονομικές κυρώσεις και τη δέσμευση των ε, στοιχείων ενεργητικού του Λουκασέγκο και των συντρόφων του. και θα πρέπει να μην λάβει χώρα στις χώρες αυτές, το, το, στη Λευκορωσία μεταξύ άλλων, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2014. Θα πρέπει να αρθεί η απόφαση αυτή και να ληφθεί άλλη απόφαση μέχρι ότου η χώρα αυτή επιδείξει ε, καλύτερη πρακτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί ο κύριος Τσπαλέκης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και πάλι να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου προς τα μέλη των ε, οικογενειών των ε, θυμάτων των ε, τρομοκρατικών επιθέσεων. Όλοι καταδικάζουμε αυτές τις επιθέσεις και καλό τις αρχές της Λευκορωσίας να εισακούσουν τη φωνή του Κοινοβουλίου και να ερευνήσουν συστηματικά τις, αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Επίσης να ανασταλούν οι εκτελέσεις των Καβάλιου και του Καναβάλιου γιατί ακόμα και τα θύματα αυτών των επιθέσεων δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη όσον αφορά την, το δίκαιο χαρακτήρα της εξαγωγής της δίκης και την, των ανακρίσεων. Η περίπτωση αυτή δείχνει και πάλι ότι δεν πρόκειται παρά μόνο για μια υπόθεση ε, χειραγωγίας και όχι επιβολής δικαιοσύνης. Εάν εκτελεστεί η θανατική ποινή, ε, θα αυξαθούν οι υποψίες ότι πρόκειται για μια άδικη δίκη. Καλό τις αρχές της ε, Ρωσίας και, άλλων, και των υπολείπων χωρών της περιοχής να καλέσουν τη Λευκορωσία να αναστείλει την εκτέλεση της θανατικής ποινής. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πελέκης. Ο κύριος Ζιάτεμάκη δεν παρίσταται, αλλά θα δώσω το λόγο στον κύριο Τσαρνέκη για ένα λεπτό. Μικρό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος Λουκασέγκο είναι μέγας ε, θαυμαστής του χόκκι στον πάγο και γι' αυτό και αρέσκεται να φωτογραφίζεται όταν επιδίδεται σε αυτή την ενασχόληση. Πιστεύω ότι θα στενοχωριόταν ιδιαιτέρως εάν το παγκόσμιο πρωτάθλημα χόκι ακυρωθεί η διοργάνωσή του στη χώρα αυτή ενώ Θα πρέπει να ασκηθεί πίεση στο Λουκασέγκο υπ' αυτή την έννοια. Και είναι πολύ σκόπιμο το γεγονός ότι συζητούμε ε, ε, το θέμα της Λευκορωσίας σήμερα είναι ένα θέμα που βγαίνει στην επιφάνεια ξανά και ξανά. Θα πρέπει λοιπόν να δηλώσουμε ξεκάθαρα ότι η χρήση μέσων όπως η, θανατική ποινή είναι κάτι το απαράδεκτο για εμάς. Και θα πρέπει να εκφράσουμε τη δυσφοδρή μας διαμαρτυρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσαρνέσκη. Ακολουθεί ο συνάδελφος κύριος Όμπερ Μάιερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Λευκορωσία είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία επιβάλλει αλλά και εκτελεί τη θανατική ποινή. Ε, παρόλο που υπέγραψαν πάρα πολλοί πολίτες ε, το έτοιμο για την κατάρριση θανατικής ποινής στη Λευκορωσία. Η τρομοκρατική επίθεση στο μετρό του Μίνσκ στις 11 Απριλίου οδήγησε στην ε, καταδίκη του Δημήτρη Καναβάλιο και του Κοβάλιοφ αλλά βεβαίως η θανατική ποινή δεν είναι η ενδεδειγμένη αντίδραση σε στη διάπραξη εγκληματικών ε, πράξεων. Και θα πρέπει οι ευρωπαϊκές χώρες να διαφοροποιούνται από τις ασιατικές και αφρικανικές παραδόσεις. Η θανατική ποινή δεν είναι δυνατόν να ε, ε, να, δεν είναι δυνατόν να, αυτή τη στιγμή έχει εκτελεστεί, δεν είναι δυνατόν να αλλάξει. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Όμπερ Μάιερ. Ο κύριος Κατσμάρεκ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι. Σήμερα συζητούμε για ένα θέμα το οποίο αποδεικνύει έμπρακτα ποιοι είναι οι κίνδυνοι που βρίσκονται γύρω από την επιβολή της θανατικής ποινής. Δεν ξέρω με ποιο κίνητρο έδρασαν οι τρομοκράτες, ωστόσο είναι σαφές ότι η θανατική ποινή είναι απάνθρωπη και μη αντιστρέψιμη. Και μάλιστα στη Λευκορωσία η θανατική ποινή δεν σταματά με την εκτέλεσή της. Το άρθρο 195 του ποινικού κώδικα στη χώρα αυτή αναφέρει ότι η οικογένεια ε, του ε, καταδικαστέντος δεν θα παραλάβει το, τη σωρό του μετά την εκτέλεση της θανατικής ποινής, ούτε καν αυτό. Απευθύνουμε έκκληση στον κύριο Λουκασένκο ε, να επιδείξει επίοικια. Είναι ένας πολύ κακός άνθρωπος και έχει τώρα την ευκαιρία να κάνει μια καλή πράξη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρέπο για ένα λεπτό. Η Λευκορωσία είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που χρησιμοποιεί ακόμα τη θανατική πίνη. Το ανώτατο δικαστήριο ε, της Λευκορωσίας αποφάσισε να, καταθήσει, ε, να καταδικάσει σε θάνατο τους ε, υπεύθυνους για την τρομοκρατική επίθεση στο μετρό του 2011. Η τρομοκρατία βεβαίω είναι κάτι το καταδικαστέο ε, που έχει σαν σκοπό να τρομοκρατήσει τον ε, πληθυσμό. Αλλά η δίκη δεν ήταν δίκαιη. Οι φυλακέ της Λευκορωσία είναι γεμάτη, ε, γεμάτες με πολιτικούς κρατουμένους. Και φαίνεται ότι οι ομολογίες αποσπώνται με την απειλή περιστρόφου στο λαιμό θα πρέπει να φροντίσουμε ε, να επιβληθούν οι κατάλληλε κυρώσει στη Λευκορωσία. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε να υποφέρει ο λαό τη χώρα αυτή. Πρέπει να τον υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρέπο. Ακολουθεί η συνάδελφος κυρία Ογιουλάντ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η εφαρμογή της θανατικής ποινής στην ουσία της είναι παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δύο καταστικαθέντες αν ήταν πραγματικά υπεύθυνοι του εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκαν, θα πρέπει να υποστούν μια ανάλογη ποινή. Αλλά δεν πρέπει να εκτελεστούν. Καλό τον πρόεδρο Λουκασέγκο να αποδώσει χάρη και στους δύο αυτού του ανθρώπου και να εφαρμόσει η Λευκορωσία μορατόριμου σε όλε τι θανατικέ ποινέ και εκτελέσει και τελικά να καταργήσει τη θανατική ποινή στη χώρα. Είναι τρομακτικό ότι ακόμα στον 21ο αιώνα υπάρχει μια ε, χώρα στην Ευρώπη που εφαρμόζει μεσαιωνικέ ποινέ. Και η Λευκορωσία πρέπει να περάσει από την ε, βυζαντινή ε, πολιταρχία στην δημοκρατική Ευρώπη ή στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά ε, την υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ογγίλαντ. Ακολουθεί ο συνάδελφος κύριος Καμίνσκι για ένα λεπτό. Ναι. Ευχαριστώ. Ε, όσον αφορά Όσο μάλλον πολιτικός και άνθρωπος, έχω όλο και μεγαλύτερες αμφιβολίες ε, σχετικά με την επιβολή της θανατικής ποινής. Αρχικά ήμουν μάλλον ε, υπέρ. Ήμουν ευνοϊκά διατεθειμένος. Αλλά σήμερα όλο και περισσότερο Είμαι ε, υπέρ αυτών που ισχυρίζονται ότι η θανατική ποινή είναι κάτι το απάνθρωπο. Αυτή είναι η μία πλευρά αυτή τη υπόθεση. Υπάρχει όμω και μια άλλη πλευρά. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για την θανατική ποινή καθ' αυτή, αλλά και για αυτό το αντιδημοκρατικό πολιτικό σύστημα. Ποτέ δεν ξέρουμε αν κάποιος έχει επιλεγεί για πολιτικούς λόγους. Ούτως ώστε το καθεστώς ε, να ε, χρησιμοποιεί τον τρόπο αυτό για να αποσπάσει την ε, προσοχή της κοινή γνώμης από τα τεράστια λάθη και λύματα και αποτυχίες του καθεστώτος. καλούμε λοιπόν να δώσει χάρη ο πρόεδρος Λουκασέγκο. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Καμίνσκι. Ακολουθεί ο κύριος Κούκαν για ένα λεπτό. Ναι, η Λευκορωσία είναι η τελευταία πολιταρχική χώρα στην Ευρώπη. Είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο το γεγονός ότι αυτή η χώρα ε, συνεχίζει να ασκεί την θανατική ποινή. Ο κύριος Λουκασένκο λέει ότι όταν παίρνει τις αποφάσεις ακούει τους πολίτες του άκουσε τους 250.000 πολίτες που υπέγραψαν ε, την, ε, το αίτημα για κατάργηση θανατικής ποινής ε, στον, στη Λευκορωσία. Η θανατική ποινή του Καναβάλιου και Καβάλιου συνοδεύεται από σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά τη χρησιμοποίηση βασανιστήριων κατά την ανάκριση. Η αθότητα των δύο αυτών ανθρώπων είναι αποδεδειγμένοι, είναι βέβαιοι. Γι' αυτό θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Λουκασέγκο να επιβάλλει ένα μορατόριο στη θανατική ποινή και να δώσει τη δυνατότητα διεξαγωγής σωστής έρευνας για τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κούκαν. Ο κύριος Μπίλαν για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο αφαίρετος χαρακτήρας της καταδίκης του Μίνσκ ε, προσέξω στις σφοδρές αντιδράσεις ολόκληρη την Ευρώπη. Τα λεγόμενα παρεκτικά στοιχεία τα οποία παρουσίασαν οι ιδιοκτικές αρχές έγιναν ε, δεκτά ε, με, συνοδεύτηκαν από σοβαρέ αμφιβολίες. Τώρα, οι εκκλήσεις για ΕΠΗ και προς τον Πρόεδρο δεν έχουν τύχει απόκρισης. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις ασφαλώς αξίζουν μια έντονη καταδίκη οι επιθέσει στο μετά του θα πρέπει επίση να καταδικαστούν. Αλλά κάθε τέτοια απόπειρα θα πρέπει να διερευνάται με προσοχή. Γι' αυτό θα ήθελα να κάνω μια έκκληση στι αρχές του Μίνσκ για μια προσεκτική ε, διεξαγωγή μιας προσεκτικής έρευνας βάσει των κανόνων που ισχύουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Η θανατική ποινή μέσω του φεκισμού του καταδικασμένου υπενθυμίζει την σταλινική περίοδο και θα πρέπει η Λευκορωσία να τηρήσει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πίλαν και τώρα ερχόμαστε στη δικασία του Catch the ε, θέλουν πάρα πολύ να πάρουν το λόγο. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Η συνάδελφος κυρία Εσάγια έχει πρώτη το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. καταδικάστηκαν οι δύο αυτοί, οι νέοι άνθρωποι λόγω διάπραξης τρομοκρατικών πράξεων. Όμως δεν ήταν μια δίκαιη δίκη. Οι παρατηρητές είπαν ότι διαπίστωσαν ότι οι κατηγορίες δεν ήταν σωστά τεκμηριωμένες και ότι ε, ε, χρησιμοποιήθηκαν βασανιστήρια κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Οι οικογένειες των καταδικασθέντων έχουν ζητήσει την ε, χάρη του Προέδρου και αν ο Πρόεδρος δεν δώσει χάρη, ανά πάσα στιγμή μπορούν να εκτελεστούν αυτοί οι δύο νέοι άνθρωποι. Ο πρόεδρος Σούλτς έχει απευθύνει διάβημα στον κύριο Λουκασέγκο να ελευθερώσει τους, ε, ε, να άρει τη θανατική ποινή Ευχαριστώ πολύ κύριε Σάια. Ο κύριος Ζόγκοφ για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ρωσία απέχει παρασάγκας από το να συγκαταλεχθεί στην κοινότητα των δημοκρατικών χωρών. Αυτό το διαπιστώνουμε στον τρόπο που λειτουργεί η δικαιοσύνη και στην ε, συνέχιση της επιβολής θανατικής ποινής. Το Συμβούλιο τέλη Ιανουαρίου αποφάσισε την εφαρμογή περαιτέρων ποινών. Ο πρόεδρος Λουκασέγκο δεν προτίθεται να αλλάξει τα πράγματα. Ενδεχομένως αξιότητες της αντιπολίτευσης θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις εξελίξεις. Ε, αποτελεί καθήκον των χωρών της Ευρώπης να στηρίξω αυτές τις δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, η Ρωσία βεβαίως μπορεί να ασκήσει πολύ μεγαλύτερη πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να κάνουμε τα αναγκαία βήματα, ούτω ώστε ο πιο στενός σύμμαχος της Λευκορωσίας αποφανθεί ότι η κατάσταση στη Λευκορωσία είναι απαράδεκτη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σόγκορ. Ακολουθεί ο συνάδελφος Γκάλαρ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Η πλειονότητα αυτού του σώματος είναι γενικά κατά της επιβολής θανατικής ποινής. Αλλά το... και το καθεστώς μας οδηγεί σε σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά τη δίκαιη διεξαγωγή της δίκης. Ο επαγγελματισμό που, με τον οποίο διεξήχθη η επίθεση στο μετρό του Μίνσκ ε, δείχνει ότι ήταν επαγγελματίες αυτοί που έκαναν την τρομοκρατική επίθεση και τέτοιου είδου επαγγελματίε βρίσκονται περισσότερο στι μυστικέ υπηρεσίε τη Λευκορωσία παρά είναι μεταξύ του πληθυσμού των πολιτών. Ε, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει μόνο να ζητήσουμε την κατάργηση θανατικής ποινή, αλλά να συζητήσουμε για την επιβολή κυρώσεων κατά του καθεστώτος της Λευκορωσίας. Ορισμένοι συνάδελφοι είπαν ίσως ότι θα έπρεπε να ακυρωθούν να ακυρωθεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα του, του χόκεϊ σε πάγο στη χώρα αυτή. Ε, για να στείλετε με τον τρόπο αυτό η κατάσταση αυτή. Συνάδελφος κύριος ε, Κέλλη έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι ομιλητές ανέφεραν ε, το γεγονός ότι η Λευκορωσία είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που επιβάλλει τη θανατική ποινή όσο ε, μέσω ποινικών ε, κυρώσεων. Από το, την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, 400 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί. 50 όμως τα τελευταία 10 χρόνια μόνο από αυτούς. Μάλλον διαφαίνεται μια ε, τάση αλλαγής στις νοοτροπίες. Ας ελπίζουμε να εξαλειφθεί τελείως η θανατική ποινή. Τώρα, ως προς τους δύο αυτούς νέους ανθρώπους, ε, αφού έχουν προκαλέσει το θάνατο τόσων πολλών ανθρώπων, αν αυτό αποδειχθεί, Σίγουρα αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο συναισθηματικό ε, φορτίο. Ε, συμφωνώ στο στην έκκληση που απευθύνεται στον πρόεδρο Λουκασέγκο να μην εφαρμόσει την απόφαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κέλλη. Η συνάδελφος κυρία Κόρολα για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως η Λευκορωσία είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που εφαρμόζει τη θανατική ποινή και αυτό είναι ένα μυστικό του κράτους. Δηλαδή οι συγγενείς, οι γονείς δεν θα γνωρίζουν ούτε την ημερομηνία ούτε τη μέρα που θα, γίνει, θα εκτελεστεί η απόφαση. Ωστόσο, έχουν καταστραφεί τα αποδεικτικά στοιχεία ε, που στήριζαν αυτή την απόφαση. Η δίκη δεν ήταν σε καμία περίπτωση δίκαιη. Θα πρέπει η Λευκορωσία λοιπόν να κάνει αληθινά βήματα προς την δημοκρατία, και προς την επικράτηση του κράτους δικαίου. Έχει έρθει πλέον η στιγμή η χώρα αυτή να ευθυγραμμίσει την νομοθεσία της με το ε, διεθνές δίκαιο το οποίο προβλέπει μια δίκαιη δίκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κόρολα. Η κυρία Τούνενστάιν έχει τελευταία το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το οποίο υπόθηκε σήμερα είναι το εξής ότι η θανατική ποινή είναι κάτι το απαράδεκτο, ανεξάρτητα από το πόσοι στην κοινωνία τίθενται υπέρ ή πόσοι κατά της θανατικής ποινής και της εκτέλεσης αυτής. Ακόμα και ο Ευρωβουλευτής ο Καμίνσκι τελικά άλλαξε γνώμη. Οι βαρβαρότητες όμως οι οποίες έχουν διαπραχθεί στη Λευκορωσία είναι κάτι το οποίο μας ε, κάνει να ε, έχουμε την υποχρέωση να αναλάβουμε πολύ συγκεκριμένες δράσεις και μάλιστα με επίγοντα χαρακτήρα. Να δεσμεύσουμε ε, την περιουσία του Λουκασέγκο, να κάνουμε το παν για να μην διοργανωθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χόκι στη χώρα αυτή, ούτω ώστε να ασκηθεί πίεση προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία έχει κλείσει η διαδικασία Catch the Eye. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Τούνουντ Χόενστάιν. Και τώρα ο επίτροπο κύριο Μπαρνιέ έχει το λόγο. Κυρίε και κύριοι, η πολυμορφία των ε, παρεμβάσεων δείχνει τις ανησυχίες ε, που υπάρχουν και τη συναισθηματική φόρτιση ε, σε όλα τα έδρανα των βουλευτών ε, μετά από τις δύο θανατικές καταδίκες του κυρίου Καναβαλόφ και του κυρίου Καβαλιόφ ε, στη Λευκορωσία. Θα ήθελα να πω εξ ονόματος της είπα της εκπροσώπου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρίας Άστον ότι μας ανησυχούν βαθύτατα αυτές οι δύο καταδίκες. Ο κύριος Καναβαλόφ και ο κύριος Καβαλιόφ καταδικάστηκαν σε θάνατο στις 30 Νοεμβρίου από τον Ανώτατο Δικαστήριο της Λευκορωσίας για την εικαζόμενη συμμετοχή του στην τρομακτική επίθεση στο μετρό του Μίνσκ το Μάρτιο του 2011 που προκάλεσε 11 νεκρούς και πάρα πολλούς ε, ε, τραυματίες καθώς και για τις τρομοκρατικές επιθέσεις το 2005 στο Βίπσκ και το 2008 στο Μίνσκ. Ε, ε, λυπούμεθα βαθύτατα για αυτή τη διπλή καταδίκη σε θάνατο. Η κυρία Άστον ε, δημοσίευσε ε, μία πολύ ξεκάθαρη δήλωση για την καταδίκη αυτής της επίθεσης, αυτής της ποινής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει, εν πάση περιπτώσει, την εφαρμογή της ανατικής ποινής. Θεωρούμε ότι πρόκειται για μία ποινή απάνθρωπη και βάναυση η θανατική ποινή δεν θα αποτρέψει μελλοντικούς ε, ε, ενόχους και είναι μια ποινή την οποία θεωρούμε απαράδεκτο όσον αφορά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κεραιότητα. Γι' αυτό ε, έχουμε δεσμευθεί για να εργαστούμε για την παγκόσμια κατάργηση θανατικής ποινή, όπω αποφασίσαμε και στου κόλπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση να την καταργήσουμε πλήρω. Με την κυρία Άστον ζητούμε από τι αρχέ τη Λευκορωσίας να μην προχωρήσουν σε εκτέλεση θανατική ποινή των κυρίων Καναβαλιόφ και Καβαλιόφα και να αναθεωρήσει την ε, θανατική ποινή. Ε, είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο που εφαρμόζει την ε, ίστατη ποινή και η θέσπιση ενό μερατόριου θα ήταν το πρώτο βήμα προς την κατάργησή της. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπαρνιέ. Ε, έχουν υποβληθεί έξι ψηφίσματα. Η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί και η ψηφοφορία θα γίνει μετά το πέρας αυτής της συζήτησης. Επόμενο, ε, επόμενη πρόταση ψηφίσματος αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις στην Αίγυπτο. Ο κύριος Μπέλντερ έχει πρώτο